Έχετε την ημερήσια διάταξη, έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή αλλαγές, όχι, εγκρίνεται λοιπόν, σημείο 2. Ήθελα να σας πω ότι υπάρχει αναμετάδοση, να μιλάτε λοιπόν αργά, ξεκάθαρα. γιατί όπως ξέρετε από το Ταλίν μέχρι τη Μεσόγειο μας κοιτούν και μας παρακολουθούν. Να σας πω επίσης ότι δεν έχουμε πορτογαλική διερμηνία. Δεν μπορείτε δηλαδή να ακούτε πορτογαλικά, αλλά μπορείτε να μιλάτε βεβαίως πορτογαλικά. Ο καθένας μπορεί να μιλάει τη μητρική του γλώσσα. Περνάω στο σημείο 3. Η κατάσταση του τριμερούς διαλόγου. Έναν τριμερή διάλογο έχουμε. Δεν βλέπω όμως τον ε, εισηγητή. Θα σας πω εγώ, πρόκειται για τον εξυγχρονισμό των μηχανισμών προστασίας των εμπορικών συναλλαγών και στην τελευταία συνάντηση που είχαμε προχωρήσαμε σημαντικά. Υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις ε, του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο μάλιστα θέλησε να αποσύρθει κάποια στιγμή. Τελικά αυτό δεν έγινε. Και υπάρχουν κάποια θέματα πολιτικά τα οποία έχουν σήμερα επιληθεί. Υπάρχει το θέμα των ε, θαλάσσιων μεταφορών, η ρήτρα για τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχει επίσης το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Εγώ την ε, Παρασκευή ήμουν στο γεύμα της TPC και έχω την εντύπωση ότι και το Συμβούλιο σήμερα είναι διατεθειμένο να προχωρήσει, να κινηθεί. Είμαστε λοιπόν πολύ πιο αισιόδοξοι σήμερα 5 Δεκεμβρίου την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η επόμενη συνάντηση και αν όλα πάνε καλά νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο στους πολίτες της Ευρώπης και στην βιομηχανία. Περνάω στο σημείο 4, μακροοικονομικές στηρίξεις. Εδώ έχουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στην έκθεση αυτή βλέπετε πολύ συγκεκριμένα αναφορές στην ε, Ουκρανία και την, ε, την Ισία θέματα αιρεσιμότητας, θέματα υλοποίησης. Όλα αυτά έχουν εξεταστεί από το ελεγκτικό συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι μπορεί τώρα να αντιδράσει. Ο Σαντιάγκο Βάκα Γκαρσία θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση του θέματος αυτού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την μικροοικονομική αυτή βοήθεια και να αναφέρουμε και τι υπόθηκε σε άλλες συναντήσεις από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου. Πρώτα απ' όλα να επενθυμίσω κάτι. Περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της χρηματοδοτήσεως αυτής. Και πώς προσεγγίζει την αιρεσιμότητα να αξιολόγηση την εποπτεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά που υπόθηκαν τότε από το ελεγκτικό συνέδριο. Να υπενθυμίσω κάτι. Αυτή η μακροοικονομική ενίσχυση είναι ένα εξαιρετικό έκτακτο μέσο σε περίπτωση ανάγκης για την αντιμετώπιση προβλήματος ισολογισμού στις χώρες της ε, ευρωπαϊκής ε, γειτονίας. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι ένα εργαλείο που κινητοποιείται κατά περίπτωση. Είναι αντίδραση σε κρίση σε εξαιρετικές και σοβαρές περιπτώσεις προβλημάτων όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών. Περιορισμένη η γεωγραφική κάλυψη. Μόνο για υποψήφιες χώρες και αυτέ που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιες χώρες στην περιοχή πολιτικής γειτονίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες που είναι γεωγραφικά και πολιτικά κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ωφεληθούν προσωρινή βραχυπρόθεσμη υποστήριξη. Η στήριξη λαμβάνει η χώρα μέχρι τη στιγμή που η χώρα θα επιστρέψει σε μια οικονομική σταθερότητα. Διαφέρει πολύ από την κανονική οικονομική υποστήριξη ή αναπτυξιακή υποστήριξη και βοήθεια. Έχει τη μορφή δανείου τυπικά. Σε κάποιες περιπτώσεις χορηγία μπορεί να δοθεί, αλλά μόνο σε δικαιολογημένες ειδικέ περιπτώσεις. Συνήθως πρόκειται περί δανείων. Χωρίς όρους. Τι σημαίνει αυτό. Οι πόροι δεν σχετίζονται με καμία συγκεκριμένη δαπάνη στις δικαιούχες χώρες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του μέσου αυτού. Στόχος είναι να βοηθηθεί δικαιούχος χώρα να αποκατασταθεί οικονομικά και χρηματοπιστωτικά και ταυτόχρονα στηρίζονται και ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Προφανώς, καλό είναι να γίνουν ιδέωσες οικονομικές προσαρμογές. Και πρέπει να εξεταστεί και ο οικονομικός αντίκτυπος των ε, προσαρμογών αυτών. Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές βασίζονται και επί συγκεκριμένης νομοθετικής διαδικασίας δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποιος κανονισμός. Κατά περίπτωση λαμβάνονται νομοθετικού περιεχομένου αποφάσεις από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βάσει προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την κανονική νομοθετική διαδικασία. Σημαντικό στοιχείο της βοηθείας. Υπόκειται σε κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα. Πολιτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ούτω ώστε να είναι επιλέξιμη μια χώρα. Τι σημαίνει αυτό. Η δικαιούχος χώρα πρέπει να σέβεται αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανικούς, να είναι ένα πολυκομματικό σύστημα το πολιτικό της, να επικρατεί το κράτος δικαίου και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι προαπαιτούμενα που ισχύουν για όλη τη διάρκεια της ε, βοήθειας. Γίνεται αξιολόγηση αν ισχύουν οι προϋποθέσεις, αν τηρούνται τα προαπαιτούμενα. Την αξιολόγηση την κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η, εξωτερική, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για όλη τη διάρκεια της βοήθειας, όχι μόνο στην αρχή. Για όλη τη διάρκεια, όπως είπα, Υπάρχει και άλλη, δεύτερη προϋπόθεση για τη χρήση του μέσου. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει πιστοτική διευθέτηση με το, ε, στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μάλλον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με συγχωρείτε, του ΔΝΤ. σε αυτό το μέσο για την οικονομική υποστήριξη οι πόροι προέρχονται μετά από, απόφαση. Είναι κοινή απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την χορήγηση τη βοηθεία. Και ανατίθεται εντολή μέσω τη αποφάσεω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί με τη δικαιούχο χώρα και τελικά καταλήγουν σε ένα μνημόνιο. Αυτό το μνημόνιο περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει η δικαιούχο χώρα, ούτω ώστε να ενισχυθεί οικονομικά και χρηματοδοτικά και να στηριχθεί η θέση της όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το μνημόνιο καθορίζει προϋποθέσεις και εκπλήρωση αυτών είναι απαραίτητη για την εκταμίευση των αντίστοιχων δόσεων. Σημαντικό λοιπόν να δούμε πώς σχεδιάζεται αυτή η αιρεσιμότητα. Καταρχάς, είναι για κάθε χώρα ξεχωριστά τα μνημόνια είναι διαφορετικά, εστάζονται επί συγκεκριμένων στόχων που θα βοηθούσαν την χώρα να αποκατασταθεί οικονομικά. Υπάρχουν διάφοροι τομείς που συμπεριλαμβάνονται, κάθε φορά όμως διαφέρουν. Θα μπορούσαν να είναι δημοσιονομική διαχείριση, χρηματοπιστωτική διαχείριση, μεταρρύθμιση του τομέα της ενέργειας, καταπολέμηση της διαφθοράς, βελτίωση του κλίματος επιχειρηματικότητας. Υπάρχει ποικιλία. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις συμφωνούνται αμοιβαίω. Σημαντικό είναι οι δικαιούχες χώρες να σπαστούν αυτά τα μέτρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να αποφύγουμε υπαναχωρήσεις και ότι δεν είναι αφοσιωμένες οι χώρες στην επίτευξη των στόχων. Εξίσου σημαντικό είναι αυτή η όρη, αυτή η αιρεσιμότητα να είναι συμπληρωματική. Πρέπει να συνοδεύεται με άλλου είδους υποστήριξη. Πιο σημαντικά χρειάζεται η στήριξη του Δούνου του και άλλα μέσα υποστήριξης ευρωπαϊκής προέλευσης όπως τα εργαλεία για τη γειτονία, εμπορικές συμφωνίες, συμφωνίες σύνδεσης κλπ. Ετοιμάζοντας λοιπόν την αιρεσιμότητα, πρέπει να δούμε πόσο συγκεκριμένα μπορεί να είναι τα μέτρα, πόσο φιλόδοξη είναι η και χρειάζεται και χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων. Σημαντικό λοιπόν να επιτευχθεί η ισορροπία. Να ακολουθείτε η μέση οδός για την αιρεσιμότητα, χωρίς να χάνουμε σε φιλοδοξία. Πρέπει να παρακολουθούνται η όροι, κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με αυτού και έχει την εξουσία να ασκεί αυτό το έργο. Η ΕΚΦΙΝ το κάνει αυτό, αλλά όχι μόνη τη και άλλε υπηρεσίε ασχολούνται με την εποπτεία. Και βασιζόμαστε και στην υποστήριξη των αντιπροσωπείων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Είμαστε ενή επαφή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Έτσι δε περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλευρά ΕΚΦΙΝ εκτελεί επιτόπιε αποστολές για να κάνει ε, επαλήθευση, εξακρίβωση. Πριν από την εκταμείευση λοιπόν της βοηθείας που μπορεί να δοθεί σε μία, δύο, τρει, τέσσερι δόσεις ανάλογα με το κάθε μνημόνιο γίνεται μια αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους. Και οι δόσεις συνδέονται με τη συμμόρφωση με τους όρους. Για να γίνει αξιολόγηση θεσπίζονται κάποιες κατηγορίες που καλύπτονται. Έχουμε κατηγορίες ε, πλήρη συμμόρφωση, μερική συμμόρφωση, δεν υπάρχει καμία συμμόρφωση και γίνεται παρακολούθηση της συμμόρφωσης της δικαιούχου χώρας με τις προδιαγραφές. Αυτοί οι όροι αξιολογούνται προσεκτικά. Λαμβάνουμε υπόψη το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα. Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Μοσκοβισή, ο Επίτροπος, περιέγραψε στην Επιτροπή τις διαφορές που υπήρχαν όσον αφορά τις δηλώσεις που έκανε και ο Σπίτσιν του ελεγκτικού συνεδρίου στη συνεδρίαση της 10 η Οκτωβρίου και για την Ουκρανία και την Τινησία πώς παρουσιάστηκαν οι ειδικές εκθέσεις. Η άποψή μας τα σχόλια των εκθέσεων όσον αφορά τα είδη των όρων και την πολιτική φύση των αποφάσεων σχημάτισε αρνητική εικόνα για τις επιχειρήσεις. Δεν υπήρχε επαρκής στήριξης από τα πορίσματα των ελεγκτών. Να τονίσουμε ότι όλες οι αποφάσεις για την Ουκρανία βασίστηκαν, όσον αφορά τη μακροοικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, βασίστηκαν στη συμμόρφωση με τους όρους. Δεν λάβαμε αποφάσεις με πολιτικά κριτήρια αποκλειστικά. Όσον αφορά το τρίτο πρόγραμμα αυτό ενίσχυσης μακροοικονομικής βοήθειας, είχαμε προβλέψει δύο εξαιρέσει για τη δεύτερη δόση. Αναφερόταν όμως σε δύο ζητήματα. για τους εσωτερικά εκτοπισμένους την αξιολόγηση και την εξαγωγή, απαγόρευση εξαγωγής εμπορευμάτων. Είχε κινηθεί δεόντως η Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε όμως ότι δεν είχαν προχωρήσει αρκετά οι προσπάθειες της Ουκρανίας. Έγινε όμως μια τρίτη εκταμείευση, μια τρίτη δόση κατόπιν ε, θέσεως άλλων δύο όρων. Έτσι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους δύο όρους για να δώσουμε τη δόση. Άλλο θέμα το οποίο σχολίασε το ελεγκτικό συνέδριο χωρίς να έχει δίκιο. Όσον αφορά τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν συνέστησε επιτάχυνση των διαδικασιών μας συνέστησε αντιθέτω, τη διερεύνηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πώ θα μπορούσε να επιταχυνθεί η διαδικασία εγκρίσεων. Απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι συστάσει τη ειδική εκθέσεω. Στείλαμε συστάσει που με τα χαρά με, τα, με δύο συνομοθετικού κλάδους να εξετάσουμε τι συστάσει. Είναι προς όφελός μας η καλή συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Έτσι τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων. Για αυτά τα εργαλεία της μακροοικονομικής ε, χρηματοοικονομικής ε, συνδρομής. Όσον αφορά τις πληροφορίες, διαβίβαση πληροφοριών, μετά από ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Επιτρόπου Μοσκοβισή και του συνσηγητού ε, Μωυσά έχουμε σημεία επαφής και έτσι υπάρχει συνεχής επαφή και διαφάνεια όσον αφορά τη βίωση πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Έτσι, στο μέλλον θα λαμβάνετε πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώματα για, για τους όρους που τίθενται για τη μακροοικονομική χρηματοπιστωτική βοήθεια. Ελπίζω ότι με αυτά που είπα να διαφώτισα κάποια στοιχεία της μακροοικονομικής αυτής χρηματοπιστωτικής αρρωγής και ελπίζω ότι στα επόμενα λεπτά θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και ενδεχόμενες, σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Έχουμε διάφορες επιχειρήσεις που αφορούν την Ουκρανία, την Ορδανία, την Τινησία και η Μολδαβία σχεδόν ξεκινά να εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Γεωργία συζητείτε για το μέλλον. Δεν έχει ληφθεί απόφαση όμως. Και ίσως να αναλάβουμε και άλλες επιχειρήσεις τέτοιου τύπου στο μέλλον. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου όσον αφορά αυτό το θέμα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας. Θα δώσω το λόγο στους αγαπητούς συναδέλφους και στον κύριο θα ξεκινήσω με τον κύριο Ίσιος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να εξηγήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, σαν εισηγητής για το θέμα της Μολδαβίας και μέλος της ΑΦΕΤ, μπορούμε να υπογράψουμε αυτές τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί η άφετε εμπλέκεται σε αυτή την συνδρομή που αφορά την μακροοικονομική βοήθεια. Η Μολδαβία δεν είναι απλώς μια τρίτη χώρα, αλλά υπάρχει συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχέσεις λοιπόν ουσιαστικά στηρίζονται σε αυτήν την συμφωνία σύνδεσης που σημαίνει στήριξη σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης της χώρας αυτής. Είναι πολύ σημαντικό η Μολδαβία βεβαίως να σεβαστεί το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του τύπου. Πέρα από αυτά τα θεμελιώδη και χωρίς την ε, αποδοχή και τον ε, σεβασμό των διαφορετικών ε, απόψεων και την έκφρασή τους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσει με επιτυχία εξευρωπαϊσμός της Μολδαβίας. Λέει ο μιλητής. Και βεβαίως εγώ θα στηρίξω πολύ θετικά κάθε πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως οι δεσμεύσεις αφορούν και τις δύο πλευρές. Κύριε Πρόεδρε, συνήθως Αυτές οι προσπάθειες οδηγούνται προς επιτυχία. Από ό,τι όμως ξέρετε, υπήρξαν προσπάθειες από μέρους της κυβέρνησης της Μολδαβίας να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Εμείς εκφράσαμε τις αμφιβολίες μας από την αρχή κιόλας, γιατί δεν είχαμε καταλάβει καλά ακριβώς τι συμβαίνει παρόλες τις ανησυχίες που εκφράσαμε και εμείς αλλά και τα κράτη-μέλη μεμονωμένα, η Μολδαβία προχώρησε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου από την αναλογική σε ένα μεικτό σύστημα. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή της Βενετίας, που είναι ένα πολύ σοβαρό όργανο υποβάλει συστάσεις εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Μολδαβία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Επιτροπή της ε, Βενετίας, λοιπόν, σε μια επίσημη ανταλλαγή απόψεων, δεν ε, κατάφερε να έχει τις ε, απαντήσεις που περίμενε. Περιμένουμε μια συνολική αξιολόγηση του νέου εκλογικού νόμου, κάτι που θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης από κοινού. Μία αξιολόγηση λοιπόν η οποία θα μας υποβληθεί όταν ολοκληρωθεί. Κύριε Πρόεδρε, προς το παρόν λοιπόν νομίζω ότι αυτή η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου του Ιουλίου του 2017 συμπεριλαμβάνει διάφορα σημεία τα οποία σήμερα ισχύουν και όλα αυτά τα σημεία συνεχίζουν να είναι επίκαιρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε που σήμερα βάλατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι ένα θέμα που έχει άμεσες πολιτικές ε, συνέπειες και διάσταση η μακροοικονομική συνδρομή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μηχανισμό και εργαλείο που διαθέτουμε για να μην απογοητεύσουμε τους πολίτες αυτών των χωρών, οι οποίοι μετά από την οικονομική ανάπτυξη περιμένουν και κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξελίξεις αυτές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρίτες χώρες με τις οποίες υπάρχουν συμφωνίες σύνδεσης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στο θέμα αυτό και το συζητάμε. Πρόκειται για ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διεθνείς συναλλαγές και θα πω ότι βέβαια το κοινό πρέπει να καταλάβει πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες, κριτήρια για το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια στα πλαίσια του πολλαετούς πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και βεβαίως και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε και ανταλλαγή απόψεων με μέλη του ελεγκτικού συνουδρίου. Θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι συναφή. Ξεκινώντας με τη Μολδαβία, θα ήθελα να πω ότι το περίφημο μνημόνιο συνεργασίας που είναι αν θέλετε η βάση για τη συνεργασία μας με την Μολδαβία γράφει ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής της συνδρομής θα πρέπει τα κράτη-μέλη να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη και απαραίτητη για την αξιολόγηση της προόδου και των διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει λοιπόν να παρέχονται εγκαίρως και με πλήρη τρόπο. Και αυτό για να αποφευχθεί κάθε είδους απάτη, διαφθορά και να διασφαλιστεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το κείμενο μας υπενθυμίζει ότι το ελεκτικό συνέδριο και με την πολύ θετική εικόνα που μας παρουσιάσατε από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αλήθεια ότι το ελεκτικό συνέδριο έδωσε τελείως διαφορετική εικόνα του τι έχει προχωρήσει. Όσον αφορά την Ουκρανία τώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας την πρόσφατη συνάντηση κορυφής της α, Ανατολικής Γειτονίας αναφέρθηκε στο 2018 και το 2019 και η κατάσταση έχει ως εξής. Επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί τα κριτήρια, πέντε από τα κριτήρια από μέρους της Ουκρανίας δεν έχουν καταβληθεί οι δόσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται τα χρήματα αυτά για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις και να πληρεί τα κριτήρια που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερεσιμότητα λοιπόν. Θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της χώρας αυτής. Και η χώρα όμως αυτή, όπως και όλες οι άλλες χώρες, θα πρέπει να πληρούν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις τους. Βέβαια, υπάρχουν διάφορες ε, φάσεις και στάδια που πρέπει να τηρούνται και να ακολουθούνται. Χρειάζονται νέοι θεσμοί για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, παραδείγματο χάρη. Τα έχουμε συζητήσει αυτά πολλές φορές. Και όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει και το θέμα της συνεισφοράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά ξέρουμε και από το ελληνικό πρόγραμμα και όλες τις συζητήσεις που είχαμε ότι πάντα ζητάμε οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες που στηρίζουμε. Αυτό λοιπόν το Μνημόνιο Συνεργασίας συνδυάζει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, κάτι που βοηθάει τους ε, πολίτες των χωρών αυτών να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας, να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και βεβαίως αυτό θα πρέπει να ισχύει και για την Τινησία και για ίσως το μέλλον ε, για τη Λιβύα. Πρέπει να στηρίξουμε τις χώρες αυτές να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Άκουσα ότι μιλήσατε για εξευρωπαϊσμό της Μολδαβίας. Ίσως δεν είναι σωστός αυτός ο όρος. Εμείς δεν θέλουμε η Τινησία να εξευρωπαϊστεί. Θέλουμε να στηρίξουμε τις χώρες αυτές έτσι ώστε να φτάσουν σε μία ανάπτυξη αυτάρκη, ανεξάρτητη και συζητήσαμε επίσης και τα ποσά τα οποία θα δώσουμε είτε σαν δάνεια είτε σαν ε, δωρεές. Ναι, με πιο αυστηρού όρου όμως και προϋποθέσεις, λέει ο Πρόεδρος. Θέλω να καλωσορίσω φοιτητέ από το Παρίσι. Καλωσορίσατε, είναι φοιτητέ ε, που εξετάζουν θέματα που αφορούν τις διεθνείς συναλλαγές στο διεθνές ε, ε, εμπόριο. Ελπίζω πραγματικά να περάσετε καλά σε αυτήν την συνεδρίασή μας, όσο μείνετε. σας άκουσα προσεκτικά. Διάβασα την ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την Ουκρανία και διαβάζω με σαφήνεια στην έκθεση αυτή ότι υπάρχουν θέματα διακυβέρνησης και υπάρχουν θέματα διαχείρισης των δημόσιων πόρων, υπάρχει θέμα καταπολέμησης της διαφθοράς που εν μέρη ήταν αποτελεσματική η δράση της κυβέρνησης αυτού τους δύο τομείς. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό δεν υλοποιήθηκε και αυτά τα σημεία που υλοποιήθηκαν δεν είναι καθόλου πιστική η υλοποίησή τους. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια. 40%, 50%, 30% υλοποίηση χρειάζεται. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της εκτίμησης. Yeah, thank Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μία προς μία στις ερωτήσεις σας. Σαφέστατα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Μολδαβία και την ε, μακροοικονομική οικονομική συνδρομή. Και αυτό το βλέπουμε και από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί γι' αυτό το θέμα. Έχουν αλλάξει οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να λάβουν υπόψη τους όλες αυτές τις επιφυλάξεις και ανησυχίες που εκφράστηκαν. Συγκεκριμένα λοιπόν το θέμα του εκλογικού νόμου. Έχει πάρει θέση η Επιτροπή ήδη. Μάλιστα υπήρξε και κοινή δήλωση μεταξύ της Αντιπροέδρου Μογκερίνη και των αρμόδιων επιτρόπων. Και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης. Πιστεύω ότι όταν ε, συντάχθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας, όλα αυτά ελήφθηκαν υπόψη και, το τελικό κείμενο τα είχε ενσωματώσει. Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας με πολύ σαφή τρόπο αναφέρει ότι έχουν ληφθεί υπόψη η κοινή δήλωση, οι αποφάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Δημοκρατία της Μολδαβίας συνυπογράφουν το κείμενο αυτό και υπάρχει αναφορά στον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, λέμε ότι όταν αξιολογηθεί τη στιγμή που θα καταβληθεί η πρώτη δόση, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα, όταν θα αποφασίσουμε για την πρώτη καταβολή της πρώτης δόσης, θα δούμε εάν πληρούνται αυτά τα πολιτικά κριτήρια και προϋποθέσεις. Και στην κοινή δήλωση λέμε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας το κατά πόσο οι αρχές της Μολδαβίας ε, λαμβάνουν υπόψη τους ε, τις ε, συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές. Υπάρχει αυτή η δύσκολη κατάσταση και όταν ε, φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση θα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εάν πληρούνται ή όχι πριν καταβληθεί η δόση. Το δεύτερο σημείο που δείξατε αφορά την Ουκρανία και το κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις είναι φιλόδοξες, είναι αποτελεσματικές και αυτό πάντα σε σχέση και με τα προαπαιτούμενα του Δουνουτού. Εδώ στο Μνημόνιο Συνεργασίας της Μολδαβίας έχει κάποιες διαφορές με την Ουκρανία. Ζητούμε πολύ φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις και στις δύο περιπτώσεις και από τις δύο χώρες. Πρέπει να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να δημιουργηθούν νέοι θεσμοί που δεν υπάρχουν και για όλα αυτά χρειάζονται κονδύλια και πόροι. Σε κάποιες περιπτώσεις, λοιπόν, Υπάρχουν κοινέ ε, προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Τομείο. Ναι, είμαστε συμπληρωματικοί στις προϋποθέσεις που θέτουμε. Το ελεγκτικό συνέδριο, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θεωρούμε το ελεγκτικό συνέδριο στα σχόλια του είναι τόσο αρνητικό στην εκτίμηση της κατάστασης. Εμείς είδαμε μια εκτίμηση σε γενικές γραμμές θετική, αναφέρθηκαν στην αποτελεσματικότητα, στην μερική αποτελεσματικότητα για κάποια από τα σχέδια αμφισβητούν η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αμφίζει τον τρόπο αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να επιδείξει περισσότερη ευελιξία Ιδιαίτερα όταν η υλοποίηση δεν είναι 100% ολοκληρωμένη. Να πει δηλαδή ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό το τομέα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Ιδιαίτερα δηλαδή όταν υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία αυτά να αναφέρονται. Αυτό λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι μάλλον σε γενικές γραμμές θετικό το πόρισμα του ελεγκτικού συνεδρίου και γίνεται αναφορά από κάποιους εδώ στην Ουκρανία σε σχέση με τις δόσεις που έχουν καταβληθεί, αναφερόμενος σε κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Κάποια σημεία δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, αλλά εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγησή μας ακόμα. Μας έχει μείνει λίγος χρόνος. Προσπαθούμε να πιέσουμε σε όλα τα επίπεδα τις αρχές της Ουκρανίας για να ολοκληρωθεί ε, η αξιολόγηση έχοντας ε, υλοποιήσει κάποιες από αυτές τις δεσμεύσεις τους. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε. Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω. Thanks a lot. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Α, ο Χέλμουτ έχει ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση που αφορά την Ουκρανία. Το τρίτο σημείο, γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, το μνημόνιο και η δεύτερη δόση καταβλήθηκε μόνο όταν είχαμε την διαβεβαίωση από το Κοινοβούλιο ότι θα περάσει νέος νόμος, το οποίο μας το υποσχέθηκαν αλλά δεν το έκαναν. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα ερωτηματικό. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει αυτή η νομοθεσία ή όχι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ε, μεταρρυθμίσεις σε αυτήν την ε, χώρα. Ξέρουμε ότι 113.000 ε, εργαζόμενοι βρίσκονται στον τομέα των δασών, στη δασοκομεία. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που αφορά τις αγορές εργασίας, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και αλλού. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για αυτό το κλάδο, στη φάση που βρισκόμαστε μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης αξιολόγησης και της καταβολής της επόμενης δόσης. Επιτροπή. Ναι, όσον αφορά τους περιορισμούς ε, για την εξαγωγή ξυλίας, μία από τις προϋποθέσεις που δεν έχουν ε, υλοποιηθεί και γι' αυτό και δεν ε, κατεβλήθη η επόμενη δόση. Υπάρχει και το θέμα των εσωτερικά μετατοπιστέντων, κάτι που δεν έχει ακόμα επίσης υλοποιηθεί, αλλά αυτό αφορά κυρίως την τρίτη δόση. Είναι προϋπόθεση για την καταβολή της τρίτης δόσης. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πρόγραμμα με τις δύο αυτές εξαιρέσεις και η φάση της αξιολόγησης που ολοκληρώνεται τώρα που ουσιαστικά προϋποθέτει περίπου τις ίδιες δεσμεύσεις και υποσχέσεις και η πίεση που ασκείται στις αρχές της Ουκρανίας για να καταβληθεί η επόμενη δόση είναι περίπου στα ίδια θέματα. Έχουν γίνει βήματα από τις αρχές της Ουκρανίας. Σε αυτούς τους τομείς ε, όμως υπάρχει στασιμότητα. Το θέμα της νομοθεσίας δεν έχει προοδεύσει καθόλου και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ε, λόγος για να μην ε, δώσουμε θετική αξιολόγηση στο σημείο αυτό. Υπάρχει επίσης και η εξαίρεση για τα προγράμματα, αν θέλετε, που αφορά αυτή η εξαίρεση. Η χρηματοδότηση έχει προχωρήσει και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες δεσμεύσεις τους. Αναφερθήκατε στο μεγάλο αριθμό εργαζομένων στον τομέα της ξυλίας, στη δασοκομεία. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς από τις συζητήσεις που είχαμε είναι ότι χρειάζονται κάποια επιπλέον μέτρα. Δεν αρκεί να συζητούμε για περιορισμούς της εξαγωγές ξυλίας και να εφαρμοστεί μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική στον τομέα αυτό στην Ουκρανία. Και υπάρχουν εδώ τρόποι και μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν στην πράξη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο. Και θα μείνουμε σε, παραμείνουμε σε επαφή όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων. Θέμα οικονομική διπλωματία. αρκετά καινοφανές ζήτημα. Ευρωπαϊκή οικονομική διπλωματία. Καμιά φορά δεν είναι ξεκάθαρο το νόημα της έκφρασης. Το έχουμε όμως το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Περιγράφει στο έγγραφο προβληματισμού για το θέμα της ε, ε, παγκοσμιοποίησης και αποτελεί ένα τμήμα της απαντήσεως προς το κοινό που θεωρεί ότι ίσως η παγκοσμιοποίηση να μην είναι επωφελής για τον απλό άνθρωπο. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσους υιοθέτησε πρόσφατα μαζί με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως περί οικονομικής διπλωματίας και είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα για τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να διαλύσετε κάπως την ομίχλη του θέματος. Και έχουμε πασίγνωστο πρόσωπο εδώ, τον κύριο Άγγελο Παγκράτη, ο οποίος είναι σύμβουλος για το θέμα αυτό της ευρωπαϊκής ε, οικονομικής πολιτικής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας καλέσατε και μου δίνετε δυνατότητα να παρουσιάσω εν συντομία την οικονομική διπλωματία, την ευρωπαϊκή και την μορφή που λαμβάνει. Με τα χαράς να είμαι ξανά εδώ στην Επιτροπή Ίντα. Μου ζητήθηκε να είμαι λακωνικός. Θα είμαι συντομότατος για να αφήσω περιθώριο για ερωτήσεις και πιστεύω θα υπάρξουν αρκετές. Αφετηρία για την κατανόηση οικονομικής διπλωματίας είναι η παγκόσμια εικόνα. Η οικονομική διπλωματία είναι κάτι που γίνεται όλο και πιο σημαντικό στον κόσμο. Για έναν απλούστατο λόγο. Κάθε χώρα στον κόσμο αισθάνεται την ανάγκη να προσαρμοστεί έναντι της μεταβαλλόμενης παγκοσμίου οικονομίας. Δεν θα περιγράψω πώς αλλάζει η παγκόσμια οικονομία. Αλλά θέλουμε να δείξουμε πώς εξηγείται αυτή η νέα φάση στην οποία περνάμε. Τα επόμενα 10-15 χρόνια 90% της παγκοσμίου αναπτύξεως θα γίνεται εκτός σύνορων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα πρέπει να συνδεθούμε με αυτή την ανάπτυξη για να διατηρήσουμε τα επίπεδα ευημερία που έχουμε. Αλλάζει η παγκόσμια οικονομία και αλλάζει ριζικά την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Έγιναν σοβαρές μελέτες και συμπεραίνουν ότι 50% από τις σημερινές της εργασίας δεν θα υπάρχουν σε 20-30 χρόνια. Και κάποιοι λένε ότι αυτό θα γίνει πιο σύντομα. Τι σημαίνουν οι αλλαγές. Ότι οι εταιρείε μας αντιμετωπίζουν πολύ σκληρό ανταγωνισμό που συνεχώς εντατικοποιείται στο παγκόσμιο προσκήνιο σε αγορές όπου η κρατική κυβέρνηση αυξάνεται και όχι το αντίθετο. Σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη στρέβλωση των συνθήκων ανταγωνισμού. Και η δύναμη της πολιτικής παίζει πιο μεγάλο ρόλο στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και θεσπίζονται κανόνες ε, που αμφισβητούνται. Και αυτό σχετίζεται με την σφαιρική εικόνα, την εικόνα για όλο τον κόσμο. Και οι πολίτες κινούνται κατά της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχει αντίδραση κατά της παγκοσμιοποίησης. Και το είδαμε αυτό και στο έγγραφο περί παγκοσμιοποίησης που αναφέρατε, Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καθορίσει το πλαίσιο και τι βασικέ έννοιε. Προσπαθούμε να το κάνουμε σε δύο εγγραφά. Η παγκόσμια στρατηγική τη κυρία Μογκερίνη, χρειαζόμαστε ισχυρή εξωτερική δράση και ο έλεγχο τη παγκοσμιοποίηση, Το άλλο έγγραφο που αναφέρατε. Στην εκμετάλλευση, στον έλεγχο τη παγκοσμιοποίησεω, αναφερόμαστε στην αυξανόμενη συνοχή των πολιτικών και των συναφών μα εργαλείων, τι κάνουμε εκτό συνόρων, στενότερη συνεργασία μεταξύ πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και εργαλείων και κρατών μελών, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και το έγγραφο ζητά πιο δραστηριοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην υποστήριξη των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στον κόσμο και ούτω τρόπο προωθώντα ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και θέλουμε να στηρίξουμε τι εταιρείε μα, κυρίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, να είναι επιτυχέστερε στο παγκόσμιο προσκήνιο. Βασικέ έννοιε δίνουν. Οι κατευθυντές γραμμές που αναφέρατε, Πρόεδρε, εκδόθηκαν τον Ιούλιο του 2017. Υπεγράφησαν όχι μόνο από το Γενικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά και από το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απευθυνόταν οι κατευθυντές γραμμές του επικεφαλής αντιπροσωπείων σε όλο τον κόσμο και απευθυνόταν και προς τις υπηρεσίες στο αρχηγείο, στις... στο κέντρο εδώ. Ε, ξεκινάμε από τις αντιπροσωπείες για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά η συνοχή είναι στα χέρια του αρχηγείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κατευθυντές γραμμές πρέπει να γίνουν κατανοητές, να θεωρηθούν πρώτο βήμα υλοποίησους, προσπάθεια να δείξουμε ότι εστιαζόμενοι επί συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και χρησιμοποιώντα τη μόχλευση που διαθέτουμε επιτυχάνουμε αποτελέσματα καλύτερα. Είναι μια κάτωθεν προσέγγισης Ζητήσαμε από όλου του επικεφαλεί αντιπροσωπείων σε όλε τι χώρε να καθορίσουν κάποιε προτεραιότητε για την οικονομική διπλωματία με σειρά προτεραιοτήτων και να προτείνουν ένα σχέδιο δράσεω για να προχωρήσουμε επί των προτεραιοτήτων. Προτεραιότητε που βέβαια θα αναθεωρούνται από την κεντρική δίκηση οι προτεραιότητε τη οικονομική διπλωματία εδράζονται επί συμπληρωματικότητα με τι ισχύουσε πολιτικέ. Είναι σημαντικότατη αφετηρία. Δεν θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική και να αλλάξουμε τι υφιστάμενε προτεραιότητε των πολιτικών μα. Θέλουμε να προσθέσουμε μια διάσταση σε σχέση με τα υφιστάμενα για να ενισχύσουμε και να συμπληρώσουμε την προσπάθεια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Υπάρχει ολόκληρο μηχανισμό, διαδικασίε που έχουν καθοριστεί σε αυτό το πρώτο στάδιο της οικονομικής διπλωματίας μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών. Θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία καταρχάς. Μιλάμε για συντομότατες εκθέσει με συγκεκριμένες δράσεις, όχι εκτενείς αναλύσεις και πολλές σελίδε αναλυτικές. Προτιμούμε εκθέσει με συγκεκριμένους στόχους και δράσει. Θα παράγουμε σαν αποτέλεσμα αυτού προτάσεις προς τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών, εκατοντάδες προτάσεις. Έχουμε πάνω από 140 αντιπροσωπείες που όλες ζητήθηκε από αυτές να καθορίσουν προτεραιότητες. Θα εξετάσουμε πολύ μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Τι θα κάνουμε τις προτεραιότητες. Ε, θα δημιουργήσουμε αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα και θα εμφανιστούν στον ιστότοπο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εμπνεύσουμε τον κόσμο. Να κινητοποιηθεί, να εστιαστεί επί των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ανάπτυξη, θέση απασχόληση, προτεραιότητα, Πρέπει να καταλάβετε ότι ήδη έχουμε εκατοντάδε μέλη του προσωπικού που έχουν κινητοποιηθεί στι αντιπροσωπείε μα και στην κεντρική δίκηση. Και αν υπολογίσουμε και τα κράτη-μέλη και κάθε χώρα στον κόσμο και τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου την άποψη ζητούμε για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, μιλάμε για μερικές χιλιάδες ανθρώπους που πρέπει να εξετάσουν το θέμα των συμφερόντων της Ευρωπαϊκή Ενώσης όσον αφορά την ανάπτυξη και θέση απασχόληση στην Ευρώπη και τον καλύτερο τρόπο δράσεως για αυτό το σκοπό. Είναι μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νοοτροπίας στη δίκηση που θα καθοδηγεί τις δράσεις μας. Χωρίς να προδικάζω τι πρόκειται να γίνει, Πρόεδρε, αυτό που είπατε για τον πολίτη είναι η ουσία. Τι προσπαθούμε να κάνουμε και τι ελπίζουμε να πετύχουμε κάποτε στα μέσα του επόμενου έτους. Έχουμε αρκετή ουσία σε αυτά που κάνουμε, ούτως ώστε μπορούμε να στραφούμε προς τους πολίτες μας, τις εταιρείες μας και τους πολίτες και να πούμε «Κοιτάξτε, σε ό,τι κάνουμε στην εξωτερική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αμελούμε τι δικέ προτεραιότητε, που είναι η ανάπτυξη και οι θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Είναι βασική προτεραιότητα για μα και για του πολίτε, βέβαια, μαζί με την ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω επί της συμπληρωματικότητα με υφιστάμενε, με ισχύσεις πολιτικέ, συμπληρωματικότητα και ενίσχυση των ισχυουσών πολιτικών, το χάρη, αναπτυξιακή πολιτική, βασικός προσανατολισμός μέσω αναπτυξιακής πολιτικής είναι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα και τους πόρους αυτού. Οι καλύτερες εκτιμήσεις για τις πιθανότητες επιτυχίας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030 προβλέπουν την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων στον αντισόμενο κόσμο. Η αναπτυξιακή πολιτική προσπαθεί να κινητοποιήσει Πόρου του ιδιωτικού τομέα να κινητοποιήσει εταιρείε να κινηθούν βάσει κοινών συμφερόντων. Αυτή είναι η οικονομική διπλωματία. Αυτό είναι ο χώρος της οικονομικής διπλωματίας και μπορούμε να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε τα όσα κάνει η αναπτυξιακή πολιτική. Όσον αφορά την εμπορική πολιτική, την ίδια αρχή ακολουθούμε. Πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο πράγματα όπως ισότιμες συνθήκες, αμοιβαιότητα, επιρροή όπου μπορούμε, χρησιμοποιώντας τους τρόπους μόχλευσης, τη μόχλευση των ανθρώπων μας για άλλου ανθρώπους, για άλλου λαού προ όφελό μας. Χρειάζεται σφαιρική προσέγγιση, παγκόσμια προσέγγιση όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής και πώς επιδιώκουμε τα συμφέροντά μας να εξασφαλίζονται. Η ε, κυρία Σάτο θα παρουσιάσει περισσότερα για τα εμπορικά θέματα. Εγώ να πω ότι η συμπληρωματικότητα ε, ενισχύει την εμπορική πολιτική. Η οικονομική διπλωματία προωθεί αυτό που πετυχαίνουμε ήδη από πλευράς εμπορικής πολιτικής για πρόσβαση στι αγορές. Δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε νέε ε, προτεραιότητες. Μπορούμε να προωθήσουμε κάποιε από τις παρούσε προτεραιότητες και συμπληρωματικότητα αφορά τον εστιαζόμεθα επί προτεραιοτήτων και συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεω που απλουστεύουν τη ζωή των άλλων γενικών διευθύνσεων και μπορούμε να βοηθήσουμε και τις δικές μας εταιρείε να κινηθούν στην παγκόσμια αγορά. Βάσει μιας πιο γενικής προσέγγισης που χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερους μοχλούς για το σκοπό. Θα αφήσω τη συνάδελφο όμως να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Είπατε ότι συμπληρώνεται την όλη εικόνα και τις προσπάθειες. Δεν αντικαθιστάται κάποιο άλλο κλάδο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς όλα αυτά εντάσσονται στην εμπορική στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συμμετοχή στη συζήτηση. Ο Άγγελος έκανε μια πλήρη επισκόπηση της οικονομικής μας πολιτικής. Εγώ να συμπληρώσω κάποια σημεία, κυρίως το πώς η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική διπλωματία. Η εμπορική πολιτική είναι βασικό στοιχείο με το οποίο ασχολείται αυτή η Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την οικονομική διπλωματία. Καταρχάς μέσω των διαπραγματεύσεων, επίσης όμως και μέσω της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών αυτό είναι κάτι άλλο που αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση των προσεγγίσεων. Αλλά έτσι συμβάλλει το εμπόριο. Επίσης, μέσω της άρσης φραγμών όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, προωθήσεως συνεργασίας όσον αφορά την οικονομική διαχείριση και διακυβέρνηση, πρόθεση ρυθμιστικής σύγκλησης και μέσω αυξήσεως της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον οικονομικό τομέα. Πράγματι, όλη αυτή η δουλειά δεν είναι καινούρια για τις αντιπροσωπίες μας και όπως και ο Άγγελος μας είπε, όλες οι υπήρες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου συνεργάστηκαν στενά, συντάσσοντας τους προσανατολισμούς που απίθυναν προς τις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το προσωπικό μας, αντιπροσωπίες τι κάνει. Ήδη ενεργά προωθούν τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξωτερικό. Οι κατευθυντήριε γραμμέ τι θα κάνουν πέραν αυτού. Θα ενισχύσουν το ρόλο των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυξήσεω του συντονισμού και μέσω αυξήσεω τη συνοχή με τι επιχειρήσει και τα κράτη-μέλη. εν παρόδο ότι διάβασα την έκθεση της Γενικής Διευθύνσεως για την Εξωτερική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οικονομική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τη σχετική στρατηγική και τι είδα. Κάτι που υπογραμμιζόταν, δηλαδή την ανάγκη στενής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και με τον επιχειρηματικό κόσμο. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω και το εξής. Αυτό είναι κάτι που ήδη κάνουμε. Πώς? μέσω των συμπράξεών μας των εταιρικών σχέσεων για πρόσβαση στις αγορές, όπου έχουμε τις αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις πρεσβείες των κρατών μελών και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που αποτελούν ένα κομμάτι της όλης δομής εκπροσώπησης σε τρίτες χώρες, και την ανακοίνωση για εμπόριο για όλους αναφέρεται στην ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων για την προώθηση των συμφερών της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο εξωτερικό. Ήδη έχουμε μια δομή, πρέπει να το πω, δεν επανεφευρίσκουμε τον τροχό, το είπε και άγγελο άλλωστε αυτό. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέε δομέ για την οικονομική διπλωματία, αλλά πραγματικά πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό και πρέπει να ενισχύσουμε τις διάφορες πολιτικές. Τώρα, όσον αφορά τον καθορισμό προτεραιοτήτων, Συλλογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντοπίσει προτεραιότητες σε σχέσεις με κάποιον εταίρο, είτε για διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, εάν έχουμε διαπραγματεύσει μια χώρα, ή για υλοποίηση, αν ήδη υπάρχει μια συμφωνία. Ή μέσω της στρατηγικής για πρόσβαση αγορές. Οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να είναι στο επίκεντρο καθορισμού προτεραιοτήτων για την οικονομική διπλωματία. Χρειάζεται συντονισμός λοιπόν για την οικονομική διπλωματία και χρησιμοποιούμε και άλλους μοχλούς, μέσα εμπορικά, Φερρυπίν. Ε, μας δημιουργούν ευκαιρίες που μπορούν να μας βοηθήσουν για την επίλυση προβλημάτων με φράγματα, με φραγμούς για πρόσβαση σε αγορές, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε αγορές, και από τις διαπραγματεύσεις ε, και διάφορα προβλήματα που απορρέουν τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο. Θέλουμε να συγκεράσουμε όλους τους φορείς, να τους συναθρήσουμε σε ένα συντονισμένο συνεκτικό πλαίσιο. Και για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Σχετικά με αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ρόλο να διαδραματίσει. Πώς, βοηθώντας να υπερασπιστούμε τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό, Νομίζω ότι εδώ μπορώ να κλείσω και με τα χαράς να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είναι πολύ καλό που ξαναβλέπουμε τον κύριο Παγκράτη να συμμετέχει στον τομέα του εμπορίου. Τον βλέπουμε σήμερα το απόγευμα. Το προσκήνιο πολύ προβληματικό πολλές προκλήσεις. Πέρα προς ανατολισμούς χρειαζόμαστε κάποιους κανονισμούς, κάποιο εργαλείο, όπου θα περιγράφονται συγκεκριμένες θέσεις, δικαιώματα και δυνατότητα να συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε αυτές τις ζυμώσεις. Είναι ένα κράμα εξωτερικής πολιτικής, ε, ε, πολιτικής εξωτερικού εμπορίου, αναπτυξιακής πολιτικής. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε αυτό το μείγμα να το αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να βρούμε και διαφανείς μεθόδους που αναλογούν στα καθήκοντά μας και τους στόχους μας. Εκτιμώ το ότι εσείς κύριε Παγκράτη αναφερθήκατε στο πρόγραμμα για το 2030 και την αναπτυξιακή βοήθεια ε, και γιατί βάσει αυτών πρέπει να αναπτύξουμε τη διπλωματία που ταιριάζουν στην παγκόσμια ευημερία και την παγκόσμια ανάπτυξη και πρέπει να προστατεύουμε και το περιβάλλον ε, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο οικονομικής ανάπτυξης που δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το υπόβαθρο. Επ' αυτού πρέπει να βασιστούμε για τις συζητήσεις. Δεύτερη πτυχή. Δεν άκουσα θεμητό, δίκαιο εμπόριο, fair trade, δεν άκουσα αυτή την έκφραση. Διότι αυτό είναι ένα τμήμα της Επιτρόπου που προωθεί η Επίτροπος η κυρία όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Και είναι μια πρόκληση για μας με σωστό τρόπο να συμμετέχουμε στο διεθνές εμπόριο. Να υπάρχει δίκαιο εμπόριο. Έχαμε διάφορες συνόδους κορυφής που έγιναν ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ONCTAD, ε, G20, Διάφοροι φορείς, διάφορα βήματα συζητούν τα ζητήματα. Υπάρχουν δομές συζητήσεων, θεσμοί και που είναι τέρι μας όλοι αυτοί οι φορείς για μια υπεύθυνη οικονομική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω τροφή προσκέψη πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη προσέγγιση. Να είμαστε διαφανείς όσον αφορά τη συνοδεία της όλης διαδικασίας που περιγράψατε. Αν μόνο 30%. Είδατε, λέει η μελέτη, 30% λοιπόν των μικρομέσων επιχειρήσεων συμβάλλουν πραγματικά στη διεθνή πτυχή των συναλλαγών και 90% της ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο παράγεται από το 30%, πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δυνατότητα να είναι κινητήρια δύναμη για δημιουργία θέσεων εργασίας. Πώς τις προσεγγίζουμε. Δεύτερη ερώτηση. Το πρωτόκολλο των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος. Πώς το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το εργοτάξιο του ΣΥΠΗΝ και δεν θα πρέπει να σκεφτούμε κοινωνικές εξελίξεις και ανάπτυξη αντί να λέμε μόνο επιχείρηση και ανάπτυξη, ανάπτυξη και βιομηχανία, να εστιαστούμε περισσότερο επί γενικότερων πτυχών όταν μιλάμε για τη διπλωματία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο ε, Ο κύριος Σένφετ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, πριν επικεντρωθώ επί του θέματός μου, θα μιλήσω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορώ να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στον κ. Σόλτς. 30% από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν άμεση συμμετοχή στις συναλλαγές εμπορικές με το εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν καθόλου, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εργάζονται για μεγάλες εταιρείες και αυτές οι μεγάλες εταιρείες εξάγουν, επανεξάγουν, όλα συνδέονται στην οικονομία. Οι πολύ μικρές εταιρείες, οι μεσές επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα και αν εργάζονται ανεξάρτητα, είναι τέτοια οικονομική κατάσταση που αφορά, απευθύνεται σε μια γενικότερη, σε, παγκόσμια αγορά. Τώρα, αυτή η οικονομική διπλωματία, πάω στο άλλο που συζητούμε μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει και το ότι τη συζητάμε σήμερα αυτή τη διπλωματία. Είναι σημαντικό θέμα, ουσιαστικό. Είναι και πολιτικό ζήτημα βέβαια. Μπαίνοντα στην ουσία. Είναι προφανέστατο ότι όταν έχουμε παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη αυτής δημιουργούν μια ενιαία οντότητα στο παιχνίδι αυτό το παγκόσμιο μέσω διαφόρων συμφωνιών τότε όλα γίνονται μέσω κυρώσεων συμφωνιών μέσω των κοινοβουλίων. Μέσω του κοινοβουλίου και όχι από τα ξεχωριστά κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι ένα σημαντικό παίκτη στο παιχνίδι αυτό. Και γι' αυτό θα πρέπει να παλέψουμε για μια κοινή οικονομική πολιτική. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο τώρα. Και θα πρέπει να το αλλάξουμε. Φυσικό είναι αυτό. Διότι τα κράτη-μέλη έχουν άλλες προτεραιότητες. Κάθε χώρα τη δική της. Διαφορετικές οικονομίες και έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς. Βιομηχανία, γεωγραφικά, έχουμε άλλες προτεραιότητες. Κάποιε χώρε ενδιαφέρει περισσότερο η Αφρική, άλλε η Αμερική, Άλλε ασχολούνται με τη βαριά βιομηχανία, άλλε με την υψηλή τεχνολογία. Υπάρχει επικοινομορφία, αλλά γενικά είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η άποψή μου που εκφράζω την πολιτική πτυχή που ανέφερα ίσως δεν πρέπει να τη συζητήσουμε εδώ. Αυτή πρέπει να συζητηθεί όμως και θα πρέπει να συζητηθεί πιο επίσημα. Γιατί και κανονιστικά είναι πιο σημαντική η πολιτική πτυχή. Και αφορά και εκείνους που πιστεύουν ότι χρειάζεται πιο μεγάλη ολοκλήρωση η Ευρώπη μια κοινή οικονομική πολιτική, η κοινή οικονομική διπλωματία. Τι μορφή θα έπρεπε να έχει στο μέλλον. Εξαρτάται κατά πολύ από το ποια μορφή θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Διότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφορά μια, μια ενωμένη Ευρώπη μια ταχύτητα, τότε έχουμε μια πολιτική. Αν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση τριών ταχυτήτων Φερρυπίν, Ευρωζώνη και η υπόλοιπη Ευρώπη και η οικονομική πολιτική, η οικονομική διπλωματία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορες ταχύτητε. Περιπλοκότατο θέμα, αλλά άκρο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν που έχουμε μπροστά μας και θα πρέπει να το συζητάμε συχνά γιατί το αξίζει. Ευχαριστώ. Ο κ. Ντάρτμουθ, συμφωνώ με τον τελευταίο μιλητή. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Πρέπει να το εξετάσουμε. Η Επίτροπος η κυρία Μάλστρομ είχε πει στην ακρόασή τη πριν γίνει επίτροπος, θα χρησιμοποιήσω την εμπορική πολιτική για να προωθήσει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα είμαι πολύ σύντομο. Προσέξτε το εξή. Συνέντευξη. Ρομπέρτο Αζεβέντο, ίσως να μην προφέρω το όνομά του. Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στη Sunday Telegraph δημοσιεύτηκε την Κυριακή. Θα μιλήσω γι' αυτό και αργότερα, σε αυτό το πλαίσιο. Παραθέτω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περικόψει περίπου 50, έχει συνάψει 50 περίπου συμφωνίες με πολύ μικρές χώρες. Παρά 60 χρόνια προσπαθειών, οι Βρυξέλλες απέτυχαν να πετύχουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία και άλλες μεγάλες οικονομίες. Γιατί, ο Ζεβέντο λέει, οι εμπορικές συμφωνίες είναι δύσκολες, αλλά υπάρχει και άλλος παράγων περιπλοκής, η γεωργία για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος εξαγωγέα αγροτικών προϊόντων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέει, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ούτω ή άλλω. Αν βάλετε από πάνω ε, στι διαπραγματεύσει για ελεύθερο εμπόριο και όλο, όλα αυτά τα τσιμπράγκαλα τη οικονομική διπλωματία, όλο αυτό το πακέτο πολιτικών στόχων, η ζωή σα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν θα πετυχαίνατε εμπορικέ συμφωνίε. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη και να το εξετάσετε παραμένει γεγονό ότι το εμπόριο ήταν η κοινή ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω από όταν είχαμε την κοινή αγορά. Και από όταν δημιουργήθηκε η ΕΚΑΧ το 1956. Το να τονίζουμε τώρα εδώ την οικονομική διπλωματία, τώρα τέτοια έμφαση στην εμπορική πολιτική μεταξύ άλλων είναι δούριο ύπο για περαιτέρω ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Και είναι αυτό που είπατε. Κάπου προδοθήκατε. Όλα αυτές οι κουβέντες, η οικονομική διπλωματία είναι ένα κομματί, ένα δομικό λίθος προ μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι το υπερκράτος. Όλα τα κράτη-μέλη ίσως να το θέλουν αυτό. Όλοι οι εκλογείς σα ίσως να το θέλουν. Αλλά ίσως και να μην το θέλουν. Και αν δεν το θέλουν, την πάθανε. Ε, έχουν εμπλέξει σε αυτό το τρένο που κάνει και πολύ θορύβο και δεν σταματάει. Ο πρέσβης, ε, αποκαλείστε εσείς ε, πρεσβευτές ο πρέσβης ήταν πολύ εύγλωτος για θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη που απαιτούνται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Οι μεσογειακές χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία, ας αφήσουμε την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες μεσογειακές στην Ευρωζώνη, η οικονομία τους χαρακτηρίζεται από χαμηλή απασχόληση, υψηλή ανεργία, πολύ υψηλή ανεργία των νέων και πολύ χαμηλή ανάπτυξη. Και αν το σκεφτείτε, αν το καλοσκεφτείτε και αν θεωρήσετε ότι η οικονομική διπλωματία θα τα θεραπεύσει όλα αυτά και όχι δραστική μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, τότε ξανασκεφτείτε το και ξανά και ξανά και πάρα πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση και από μένα. Βεβαίως, νομίζω ότι είναι λογικό να σταθεροποιηθεί η οικονομική ανάπτυξη βάσει των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά το επόμενο ερώτημα είναι ποιος μπορεί να ορίσει ποια είναι τα συμφέροντα τα ευρωπαϊκά. Διότι έχουμε διαφορετικά κράτη-μέλη, διαφορετικές πολιτικές προοπτικές και όλα αυτά καθιστούν ε, κολύπλοκο ένα σωστό ορισμό. Όσον αφορά το ερώτημα του Χέλμοντ. Βεβαίως, έχουμε εδώ πολλούς εμπλεκόμενους οι οποίοι προσπαθούν ε, να σταθεροποιήσουν τα οικονομικά, όπως το G20. Ποια είναι η σχέση μεταξύ όλων αυτών. Υπάρχουν κάποιες κοινέ απόψεις στα πλαίσια αυτής της οικονομικής διπλωματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τις πολύ απλές αυτές ερωτήσεις. Πολύ προκλητικές, δεδομένου ότι αναφέρονται σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να ξεκινήσουμε από εδώ. Βασικά, όμως, το, η βασική απάντηση στα ερωτήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων του κυρίου Ντάρτμουτ, δόκτωρο, πώς να σας αποκαλέσω. Ξιότιμε, κύριε Ντάφμον; Αυτό λοιπόν το οποίο κατά την άποψή μου είναι πρωταρχική σημασία στα πλαίσια της οικονομικής διπλωματίας για να ανταποκριθούμε σε αυτά τα μελήματα και τα ερωτηματικά στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενσωμάτωση έχουμε όλοι θεμελιώδου σημασία καθήκον και συμφέρον και καθήκον προς τους πολίτες μας να τους παράσχουμε τα κοινά αγαθά τα οποία δεν μπορέσαμε με τα ήδη υπάρχοντα μέσα που έχουμε στα χέρια μας. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, δηλαδή Προσπαθούμε να δούμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο που να γίνει αποδεκτό και να καθορίζεται για σε ειδικά θέματα από όλους τους πολίτες μας. Η προσέγγιση η δική μας προς τις αντιπροσωπείες και τους επικεφαλείς των αντιπροσωπειών και τα, ε, οι εκθέσεις που θα ασχολούνται με το θέμα αυτό είναι ότι αν υπάρχει ένα κράτο μέλος το οποίο ε, δεν ε, συμφωνεί ή έχει τρομερές αμφιβολίες και αμφισβητήσεις για μία από τις προτεραιότητες να μην τις συμπεριλάβουμε στον κατάλογό μας, διότι χρειαζόμαστε την πραγματική ε, βοήθεια και προσπάθεια εκ μέρους όλων των επικεφαλής και πρέσβεών μας. Θα πρέπει να είναι όλοι σε θέση να καθορίσουν έναν σημαντικό αριθμό προτεραιοτήτων με τις οποίες συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη και συμφωνούν ότι πρόκειται για κοινό συμφέρον, συμφέρον όλων των πολιτών για να προσπαθήσουν να τις προωθήσουν όπως μπορούν. Και αυτό είναι θέμα ευθύνης στα πλαίσια της παρούσας κατάστασης της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. Αυτό απαντά επίσης και τον ε, ερώτημά σας, Πρόεδρε. Ποιος το καθορίζει. Αυτή τη στιγμή η προσέγγιση μας είναι από τη βάση προς τα πάνω διότι οι προτεραιότητες πρώτα απ' όλα καθορίζονται από τους πρέσβους μας από κάτω, όπως σας είπα, με αυτή την προοπτική, με αυτή την προσέγγιση, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία πέρι αυτών και για το γεγονός ότι θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία για όλα τα κράτη-μέλη μας. Η οικονομική διπλωματία έτσι όπως ορίζεται σήμερα. Δεν ξέρω τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, θα το δούμε. Αλλά δεν προβλέπω το μέλλον. Λέγω έτσι όπως ορίζεται σήμερα. Δεν επηρεάζει την ικανότητα που έχουμε να κάνουμε συμφωνίες τώρα ή στο μέλλον. Δεν είναι απευθείας μέρος των διαπραγματεύσεων που θα κάνουμε για τις περαιτέρω συμφωνίες. Οι προτεραιότητες είναι επιχειρησιακές, λειτουργικές, δηλαδή πρακτικά βήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και πιστεύουμε ότι αν ενεργήσουμε από κοινού με τα παρόντα μέσα που έχουμε και με τις τους παρόντες πόρους μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα προς όφελος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, το γεγονός ότι δεν έχουμε συμφωνίες με τους πρωταγωνιστές του εμπορίου, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν ε, παγκοσμίες τέτοιου είδους συμφωνίες. Πρόκειται για μία μεγάλη πρόκληση για όλους, για όλους λέγω γενικότερα. Οι σχέσεις με το G20 και άλλους φορείς. Σκεφτείτε αυτά τα οποία είπαμε για την ε, συμπληρωματικότητα. Δεν επηρεάζουμε το πλαίσιο των παρουσών πολιτικών. Προσπαθούμε να βρούμε συμπληρωματικά θέματα τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις μας να είναι πιο ανταγωνιστικές, πιο προορατικές, αλλά δεν επηρεάζουμε την κατάσταση έτσι όπως έχει Μιλούμε για συμπληρωματικότητα, που είναι στοιχείο κλειδί για να καθορίσουμε τις προτεραιότητάς μας. Ζητούμε τις πρέσβεις μας ανά τον κόσμο, μαζί με τις πρεσβείες των κρατών μελών, να κάνουν οτιδήποτε μπορούν ώστε να θεωρηθούν ως προτεραιότητες της οικονομικής διπολβετσίας και όλα αυτά τα θέματα να περάσουν από τις Βρυξέλλες και εμείς θα τα βοηθήσουμε, θα τα προωθήσουμε και θα βοηθήσουμε και όλες τις προτεραιότητες. Προσπαθούμε λοιπόν αυτό το στοιχείο της συμπληρωματικότητας να το έχουμε κατά νου και αυτό είναι και θέμα που αφορά τις προτεραιότητες που παίρνουν και στα, παίρνουν και στα πλαίσια του G20 Φερρυπίν. Τώρα, όσον αφορά το επιχειρήμα του κυρίου Σόλτς, η Fairtrade, το δίκαιο εμπόριο, όντως, λείπει ο όρος. Αλλά Περιφραστικά τα είπαμε αυτά και η συνάδελφος και εγώ. Όλα αυτά τα θέματα. Σε όλα τους τομείς που αναφέραμε το λαμβάνουμε υπόψη. Και συμφωνώ με ό,τι είπατε για το ε, Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, για την κοινωνική ανάπτυξη, για τις προσπάθειες συμπληρωματικότητας των πολιτικών που ακολουθούνται σήμερα, βάσει των αξιών μας. Βεβαίως, δεν θα κάνουμε εις βάρος των ε, αρχών και των αξιών μας κάτι στα πλαίσια της ε, οικονομικής διπλωματίας. Συμπληρωματικά ενεργούμε, όπως σας είδα. Αυτή είναι η προσέγγιση μας και στην εμπορική πολιτική και σε άλλες. Δεν υπάρχει καμία αντίθεση. Προσπαθούμε από κοινού να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των στόχων μας βάσει των αξιών μας. Το θέμα των ε, ΜΜΕ και του διεθνούς τους ρόλου. Αναφέρθηκε δύο φορέ το θέμα αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τον κύριο στόχο των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ε, θα κάνουμε κάτι το επαναστατικό για να υποστηρίξουμε την διατνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αύριο το πρωί, αλλά βεβαίως πρόκειται για ένα από τα μεγάλα μελήματα της οικονομικής διπλωματίας. Έχουμε αρχίσει να κάνουμε επιτυχή βήματα Έχουμε πρώτα απ' όλα κάποιον κατάλογο των μέσων που διατίθενται για να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μιμιέ σε όλες τις χώρες μας και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να τις βοηθήσουμε. Φερρυπίν να πληρώσουμε κάποια κενά. να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία αρχίζει τώρα να τίθεται σε εφαρμογή, αλλά η υποστήριξη η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι από τα μεγάλα μας μελήματα. Τώρα, σε σχέση με τα κλιματική αλλαγή και το πρωτόκολλο του Παρισιού. είμαστε σε διαδικασία ανάπτυξης του τι σημαίνει αυτό στην πρακτική. Προσπαθούμε να ορίσουμε για κάθε σημαντικό θέμα στα πλαίσια της κάθε αρμόδιας γενικής διεύθυνσης πώς όλο η μηχανή για την οικονομική διπλωματία μπορεί να τεθεί συγχρονισμένα σε εκκίνηση. Και βεβαίως και βλέπουμε και ποια είναι και ο συντονισμός όλος αυτός και η προκλήση που στα πλαίσια γενικότερα της υποπλατείας της κάθε χώρας. Οτιδήποτε κάνουμε έχει ως στόχο την αηφόρο ανάπτυξη. Δηλαδή, προσπαθούμε αυτή να είναι η στόχη μας για όλους και όχι μόνο για την αναπτυσσόμενο κόσμο. Η στόχη μας στα πλαίσια λοιπόν της οικονομικής διπλωματίας αφορούν όλες τις χώρες. Το θέμα που έφερε ο κύριος Τζένσφελ και συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Όντως, από πολιτικής και οικονομικής πλευράς συμφωνώ και αυτός είναι ο στόχος ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια κοινή οικονομική πολιτική πέραν των συνόρων μας. Σωστά το θέσατε, συμφωνώ. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Βεβαίως όλα εξαρτώνται από τι θα είναι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όπως είπα είμαι πεπισμένος ότι έχουμε ακόμη μεγάλο περιθώριο ελιγμό να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον κόσμο και στους πολίτες μας. Κατά πρώτο λόγο. Βεβαίως, έχουμε προβλήματα. Βεβαίως, πολλοί ενεργούν και στα πλαίσια των πολιτικών μας μέσα σε στεγανά. Θα πρέπει λοιπόν να άρουμε τα εμπόδια και να ενεργήσουμε με τρόπο που θα είναι επωφελής για όλους τους πολίτες μας. Αυτός θα πρέπει να είναι, αυτή θα πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη και πιστεύω ότι όσο προχωρούμε σε αυτή τη συζήτηση, ο ρόλος που θα διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σημαντικός. Διότι έτσι μπορούμε με πρακτικό και λειτουργικό τρόπο να προσεγγίσουμε περισσότερους πολίτες χωρίς να δημιουργήσουμε ένα υπερκράτος Μπορεί να χρειαζόμαστε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα υπερκράτος για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Διότι σας είπα, έχουμε περιθώριο ελιγμών και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστώ. Δεν είναι απαραίτητο το υπερκράτος. Ένα είναι αρκετό. Uh, uh, um, Κυρία Ράτσε, όπως είπε ο Άγγελος με πολύ λεπτομεριακό τρόπο, και που εφόσον είπε τα πάντα δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά. Ξέρω ότι πολλά μέλη τη Επιτροπή σα ενδιαφέρονται για το πώ μπορούμε να προωθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Α πω λοιπόν κάποια πράγματα, γιατί ο κ. Σένφιλ και ο κ. Σόλτ ανέφεραν αυτή τη διάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρώτα απ' όλα, ακόμη και αν πρόκειται για 13% των ΜΜΕ, που είναι διεθνείς, δηλαδή εξάγουν εκτός ευρώ, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κλασικό παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι αρχίζουν να διεθνοποιούνται οι διεθνείς, σε διεθνές επίπεδο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτα απ' όλα εκτείνονται στις γειτονικέ τους χώρες και μετά αρχίζουν να εξάγουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. 25% των εξαγωγικών εταιριών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μιμιέ. Τι σημαίνει ότι η πλειοψηφία των εξαγωγέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, το ίδιο ισχύει με την οικονομική και στην οικονομική διπλωματία. Αυτοί που ωφελούνται περισσότερο είναι οι ΜΜΕ, διότι οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να αντεπεξέλθουν και στους φραγμούς που τίθενται από τις διάφορες ε, διεθνείς αγορές. Έχουν ε, πολύ ισχυρές νομικές υπηρεσίες, έχουν χρήμα, αλλά οι μιμιέ που επωφελούνται περισσότερο είναι οι μικρές. Και βεβαίως αυτό το οποίο λείπει ο ρησός είναι η συμπληρωματικότητα. Αυτό το οποίο κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέρη είναι να συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την προώθηση των εξαγωγών και για την προσέλκυση επενδύσεων για τις χώρες αυτές. Παρ' όλα αυτά, όταν έχει κανείς να αντιμετωπίσει διαφορετικές αγορές και διαφορετικά προσκόμματα, δεν είναι σε θέση ούτε κάθε χώρα χωριστά. Ίσως μπορεί να είναι αυτή η θέση της Γερμανίας ή την ε, ε, Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν ε, ισχυρές πρεσβείες στο εξωτερικό. Υπάρχουν όμως χώρες που δεν διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή. υποδομή. Άρα, εάν κάνουμε την κατάλληλη δράση και έχουμε την κατάλληλη στρατηγική και βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε πάρα πολύ αυτές τις εξαγωγικές μιμιέ και αν έχουμε και την ε, υλοποίηση κοινών στόχων, μπορούμε να θέσουμε όλους τους πόρους που διαθέτουμε από κοινού για να αυξήσουμε τις δυνατότητες των μήμων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, λεπτομερείς πληροφορίες που μας δώσατε και είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή μας θα είναι στο πλευρό σας και θα σας συμβουλεύει όταν χρειάζεται.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 ask first the coordinators of the political groups and then the other members to raise remarks, questions, criticism, or whatever they want. Joseph. Thank you very much, Chairman. Um, yeah, it's a pleasure to be here again. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη ευχαρίστηση είμαι εδώ. Είχα έρθει πριν από μερικές εβδομάδες, τώρα έχω περισσότερο χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με την έκθεση αυτή το οποίο περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες. Πρόκειται για ανακοίνωση, για έκθεση η οποία περιέχει πληροφορίες ανα τομέα, περιοχή, ένα χώρα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά τα θέματα τα οποία θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας. Είναι σαφές ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι θα έχουμε τις πρώτες σας αντιδράσεις και να δούμε όλοι συλλογικά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρόκειται για ένα σχέδιο που άρχισε φέτος. Ανακοινώθηκε από την Επιτροπή με χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από όλε τι υπηρεσίε τη Εμπλεκόμενη Επιτροπή να συντάξουν την έκθεση. Πρόκειται για μια πρώτη έκθεση, θα θέλαμε να γίνει αιτήσια και να τη χρησιμοποιήσουμε. Όχι μόνο για να τη δημοσιεύσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, δεδομένου ότι έχουν ε, θετικό αντίκτυπο στο εμπόριο, σε εμπορικέ συναλλαγές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θέματα τα οποία μας ανησύχουμε, τα PUR, τα θέματα των προτιμήσεων, Πράγμα που σημαίνει ότι οι διάφορες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν την δυναμικότητα που μπορούν να έχουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτή είναι η πρώτη μου σημαντική παρατήρηση. Έχουμε κάποιες ιδέες για το τι συμβαίνει, για, τι, για ποιο λόγο συμβαίνουν τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε αποφάσεις όπως ξέρουμε. Εάν δείτε τους διάφορους τομείς που εφοβελούνται περισσότερο σύμφωνα με τα δεδομένα είναι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας και η γεωργία. Η γεωργία είναι πολύ ενδιαφέρον τομέας δεδομένου ότι και στα μέσα και με ε, τις διάφορες πολιτικές μας η γεωργία θεωρείται για ε, πολλού αμφιλεγόμενου τομεί παρά το γεγονό ότι είμαστε για γεωρικά προϊόντα ω Ευρωπαϊκή Ένωση οι μεγαλύτερο εξαγωγέ παγκοσμίω. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό. Ξέρω ότι η Επιτροπή σα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα είναι πάρα πολύ υπέρ τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, υπάρχουν ειδικά κεφάλαια αφιερωμένα στο θέμα αυτό. Όπω σα είπα, βρισκόμαστε ακόμη στην εκκίνηση όσον αφορά τις συμφωνίες εμπορίου. Είμαστε ακόμη λοιπόν στην αρχή, στο α, αλλά πρέπει σιγά σιγά να προχωρήσουμε από κοινού. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά και βεβαίως με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τις ερωτήσεις των συναδέλφων και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. God live εκ μέρους του ΕΛΚ. Μιλώ εξ ονόματος της συναδέλφου η οποία είναι στο Παρίσι γιατί ιδρύεται ένα καινούριο κόμμα, δεν είναι εδώ. Και είναι αρμόδια για αυτό το θέμα. Και δεν θα μιλήσω αγγλικά, θα μιλήσω γαλλικά. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή και τη μελετούμε προσεκτικά στα πλαίσια της σύνταξης σχεδίου ψηφίσματος για την ευρωπαϊκή ε, εμπορική πολιτική. Είναι λοιπόν απαραίτητο να κάνουμε μία περιστατωμένη ανάλυση της εμπορικής πολιτικής. Θα ήθελα να επιμείνω σε πολλά σημεία και να υποβάλω ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, γενικά, από τις διάφορες συμφωνίες βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικοί αριθμοί, πράγμα που αποδεικνύει ποια είναι τα ωφέλη από τις ε, ε, συμφωνίες αυτές και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί δεν γίνονται αυτά περισσότερο γνωστά, δεν είναι περισσότερο γνωστά. Πάντα μιλούμε για κινδύνους, για ρίσκα, αλλά λιγότερο για τα θετικά σημεία και τα πλεονεκτήματα. Όσον αφορά την χρησιμοποίηση των εμπορικών προτιμήσεων, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λιγότερο τα ωφέλη, παρότι οι επιχειρήσεις των ε, εταίρων χωρών. Μπορείτε να μας πείτε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ποιοι είναι οι λόγοι. Τι είδους δράσεις θα κάνετε για να μπορέσετε να διορθώσετε αυτή την κατάσταση. Ποια είναι τα μέσα τα οποία θέτουν, θητίθενται σε εφαρμογή στις χώρες εταίρους που καταλήγουν στο να χρησιμοποιούν περισσότερο και καλύτερα τα ωφέλη από αυτές τις συμφωνίες. Τρίτον, στα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής αναγγέλει η Επιτροπή την δημιουργία οδικού χαρτί για τις συμφωνίες αυτές. Πρόκειται για ένα μέσο πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο θα είναι και χρήσιμο για να παρακολουθήσουμε και πώς τίθεται σε εφαρμογή συγκεκριμένα κάθε τέτοιου είδους συμφωνία. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ε, πληροφορίες για αυτό τον οδικό χάρτη και με ποιο τρόπο θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί. Τέταρτη ερώτηση. Ένα σημαντικό σημείο που για μας τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους είναι πρωταρχική σημασία. Ποιος είναι ο ρόλος των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντιπροσωπίες είναι σε άμεση σχέση με τους οικονομικούς φορείς επιτόπου, με την ε, κοινωνία των πολιτών και με τις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες βρίσκονται. Θα πρέπει λοιπόν να τι υποστηρίξουμε και να συγκεράσουμε τις δράσεις τους με τις δράσεις των αντιστοίχων αντιπροσωπιών στις χώρες εταίρους. Τελευταία παρατήρηση. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται και δύο θέματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένω να μας ανησυχήσουν. Πάντα σχεδόν τα ίδια. Πρώτα απ' όλα, η πρόσβαση στις δημόσιες αγορές και δεύτερον η προστασία των ΠΟΠ στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Ως ΕΛΚ πάντα είμαστε υπέρ αυτών των δύο διαφορετικών στοιχείων, αλλά πολλές φορές αναφέρεται ότι υπάρχουν προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν σε κάποιες συμφωνίες και οι διατάξεις που προβλέπονται δεν γίνονται πάντα σεβαστές. Είναι λοιπόν πρωτορχική σημασία να παρέμβουμε για να βρούμε λύσεις. Εξάλλου για τις δημόσιες αγορές, για τις κρατικές προμήθειες θα πρέπει να ξέρουμε χάρη στη συμφωνία πόσο άνοιγμα δίδεται και να έχουμε καλύτερη επικοινωνία σε αυτό το είδος τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε για τις παρεμβάσεις σας. Όπως γνωρίζετε ζητήσαμε επανειλημμένα να γίνει εμβάθυνση όσον αφορά την υλοποίηση των μέτρων που είναι σημαντικό κομμάτι όλης της διαδικασίας ολοκληρώσεων των διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή που ψηφίζεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι σημαντικό, πιο σημαντικό να αξιολογηθούν οι εξελίξεις και η εφαρμογή της συμφωνίας. Και εγώ έχω κάποια σημεία, κάποια αναφέρθηκαν ήδη από τους συναδέλφους, αλλά επαναλαμβάνω διότι πιστεύω ότι και από την πλευρά μας είναι σημαντικό να έχουμε κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μας, είναι θεμελιώδη σημασία να κατανοήσουμε ποια είναι τα εργαλεία για να κοινοποιούμε καλύτερα τα αποτελέσματα, να τα προβάλλουμε από τα αποτελέσματα των εκθέσεων, να τονίζονται, διότι ζήσαμε και ζούμε αυτή την περίοδο μια συζήτηση στρεβλή σε σχέση με την έλλειψη στοιχείων περισσότερο βασίζονται σε αντιλήψεις παρά σε στοιχεία. Για μας είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να διαδώσουμε τα αποτελέσματα καλύτερα και να διαθέτουμε τα στοιχεία στην κοινή γνώμη. Και αυτό αφορά ένα μεγάλο τμήμα των εργασιών του Κοινοβουλίου, Της προσπάθειας που να κάνει το Κοινοβούλιο, να προβάλλει τον δημοκρατικό έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιούμε και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε. Δεύτερο, και αυτό αναφέρθηκε. Σημειώσαμε και εμείς ότι υπάρχει δυσανάλογη χρήση των εργαλείων αυτών, των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, κυρίως από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, έναντι των ομολόγων μας. Είναι θέμα επικοινωνίας αυτό. Θέμα διάδοσης πληροφοριών. Και πώς να φροντίσουμε να συμμετέχουν πιο πριν και περισσότερο οι εταιρείε, ώστε τα αποτελέσματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι καλύτερα και πιο ομοιογενή. Τρίτο. Τον οδικό χάρτη εφαρμογή, Implementation Roadmap. Πώς προτίθεστε να προχωρήσετε στο μέλλον, Βάσει αυτού, τι θα είναι, κάποιο έγγραφο, κάτι που θα προσαρτάται στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που θα εξελογεί το Κοινοβούλιο. Τεχνικός πώς. Πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε, να κινηθούμε όσον αφορά τους οδικούς χάρτες. Αναφερθήκατε στο κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, αηφόρου αναπτύξεως, sustainable development. Μας ενδιαφέρει πολύ. Πιο συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να πετύχει την έγκριση πιλωτικού προγράμματος σχετικά με τη συλλογή μη ομαδοποιημένων στοιχείων. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, τις συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών, τι αντίκτυπο έχουν οι συμφωνίες, περισσότερα ωφέλη, λιγότερα ωφέλη, όσον αφορά την οικονομία σε σχέση με τις γυναίκες. Μπορούν αυτά τα στοιχεία για να ολοκληρώσουμε τις εκθέσεις στο μέλλον και τη γενικότερη εικόνα. Αυτά και ευχαριστώ. Ehm, Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω, διότι πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά είχαμε τέτοια ενημέρωση όσον αφορά αυτούς τις διαφορετικές συμφωνίες που συνάπτουμε με τρίτες χώρες και σε όλες τις φάσεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο Φερρυπίν θα πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει πάντα να ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος κάποιων διμερών ε, συμφωνιών σε σχέση με άλλες. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν και την οικονομία και την κοινωνική ε, πραγματικότητα των κρατών μας και εδώ και σε επίπεδο των εταίρων μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο οι συνάδελφοι που είπαν ότι είναι καλό αυτό διότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ε, ευαισθητοποιήσουμε και διάφορους, ε, ε, διάφορα άτομα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα είναι σωστό. Θα ήθελα όμως να πω ότι εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει επίσης είναι τα κριτήρια. Ποια είναι η συγκριτική ανάλυση που έχει γίνει για να δούμε πώς ε, ε, λειτουργούν τελικά αυτού του είδους οι συμφωνίες. Προηγουμένως στις συζητήσεις που είχαμε για την ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και την οικονομική διπλωματία. Είπαμε επίσης ότι το benchmarking, αυτή η συγκριτική ανάλυση είναι χρήσιμη και για να δούμε πώς θα προωθήσουμε τις εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να δούμε πώς έχει και η ανάπτυξη στις χώρες με τις οποίες συνάπτουμε τέτοιου είδους συμφωνίες. Δεν θα πρέπει λοιπόν πάντα να προσπαθούμε σε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες και συναλλαγές να προσβλέπουμε σε μια ισόρροπη κατάσταση. Στην σελίδα 31 μιλούμε για το Μεξικό, την καταπολέμηση φτώχεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις ανισότητες και λέγεται ότι οι συμφωνίες της ΕΦΤΑ δεν έχουν καμία επίπτωση. Αν εξαφανιστεί ο γαλακτοκομικός τομέας δεν θα έχουμε αντίκτυπο στην απασχόληση ή στην ε, ύπεθρο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν μέχρι πού φτάνει ο αντίκτυπος όλων αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Όταν οι εισαγωγές μας από την Κολομβία μειώθηκαν από τότε που υπάρχουν τέτοιου είδους συμφωνίες κατά 37% μελετήσαμε τι συμβαίνει. Ποιοι είναι οι τομείς που υποφέρουν από αυτό τον μείωση και τον αντίπτυκο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε όλοι από κοινού να σκεφτόμαστε αυτό πράγματα για να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μετρήσουμε τον αντίκτυπο και να καθορίσουμε τα κτηριτήρια για αυτού του είδους τις εμπορικές συναλλαγές δεδομένου ότι είναι σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι βεβαίως πρέπει να παρακολουθούμε και τις πολιτικές εξελίξεις και να δούμε τι μελλοντικές ε, στρατηγικές ε, θα αναπτύξουμε. Παραδείγματο χάρη για την ε, Μπελαρούς. Μιλάμε για το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος μας στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών. Και βεβαίως είμαστε ένας οικονομικός εταίρος, αλλά στην πράξη υπάρχουν και άλλα θέματα που μας απασχολούν. Στην Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της υλοποίησης μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και το θέμα της πολιτικής αξιολόγησης που συμβαδίζει πόσο λένε τα δεμένα είναι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εγώ δεν διαβάζω τα πράγματα όπως εσείς και διαφωνώ όσον αφορά αυτά που είπατε για το αγροτικό τμήμα αυτής της συμφωνίας και πιστεύω ότι με την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας θα υπάρξει μεγάλη πίεση στον προϋπολογισμό. Έχουμε αξιολογήσει τον προϋπολογισμό για το 2019-2024 όσον αφορά τα αγροτικά θέματα που σήμερα είναι 460 δις ευρώ θα μειωθούν κατά 60 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την ε, γεωργία. Και δεν νομίζω ότι οι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου θα καλύψουν αυτό το κενό, κυρίως όσον αφορά τη συνοχή. Οι πιο δυνατές χώρες στον τομέα της γεωργίας είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Αν προσθέσουμε εδώ και τα θέματα που γνωρίζουμε στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελεύθερου με το Μερκοσούρ, τα πράγματα επιδεινώνονται. Δεν λαμβάνετε κατά τη γνώμη μου λοιπόν σωστά όλες αυτές τις συνέπειες της αξιολογής σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Κόρκου, για την παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να γνωρίσω ότι όντω η Επιτροπή εστιάζεται στην σημασία αυτού του είδους των εμπορικών συμφωνιών, δεδομένου ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό. Σέβομαι τις προτάσεις που θα μπορούσαν ε, να βελτιώσουν την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία διαφοροποίηση ως εξή. Τι μεταξύ δηλαδή εφαρμογής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χώρες εκτός. Όσον αφορά το τι συμβαίνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να έχουμε μία σωστή στρατηγική επικοινωνίας για το τι σημαίνουν όλες αυτές οι συμφωνίες. Πολλές φορές ε, έρχομαι σε επαφή με άτομα του τομέα των επιχειρήσεων και δεν γνωρίζουν σχεδόν καθόλου περί τίνος πρόκειται. Τουλάχιστον στην αρχή της περίοδου διαπραγμάτευσης μπορεί να υπάρχει ενημέρωση, αλλά μετά υπάρχει ε, άγνοια ενημέρωσης με απλό τρόπο για το τι συμβαίνει. Και αυτό είναι κάτι που είναι χρήσιμο για τις επιχειρήσεις. Είναι σωστό μέσο η ιστοσελίδα της Επιτροπής, αλλά ήθελα να ξέρω ποιο ποσοστό πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οι ΜΜΕ, κυρίως για να υποφεληθούν. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την προσπάθεια εκ μέρους των κρατών μελών. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάποιο έλλειμμα και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για εμπορικά θέματα, αλλά για την προώθηση υπάρχει κάποιο κενό. Όσον αφορά τρίτες χώρες, νομίζω ότι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, κυρίως για αυτές θα μιλήσω πρώτα, ε, δεν έχουν εκ μέρους μας τον κατάλληλο σχεδιασμό εφαρμογής τέτοιου είδους συμφωνιών. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το λάβετε υπόψη. Εγώ έφτασα το πριν από λίγο από την Κεντρική Αμερική, στην Κοσταρίκα, που και εκεί μπόρεσα να συναντήσω διάφορους φορείς, επιχειρηματίες, α, μη, ε, ε, κοιό και τα λοιπά. Και μου είπαν το ίδιο η δομή τους η επιχειρησιακή, που δεν σημαίνει ότι δεν έχουν θεσμικό πλαίσιο στη χώρα τους, δεν μπορούν να εφαρμόσουν το σύνολο των κανόνων των ευρωπαϊκών. Πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Εάν αυτές οι μιμίε δεν έχουν τις ηθίκες που θα τους επιτρέπουν να πληρούν τους κανόνες και τα στάνταρ μας, όσο καλές και να είναι οι προθέσεις τους, όσο και οι ωραίες συμφωνίες προτιμησιακές έχουμε, δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τους κανόνες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κάποια θέματα τα οποία προβλέπονται για την άρση κάποιων εμπορίων για ακόμη και για θέματα τελών που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και σε χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής και σε άλλες χώρες πρέπει να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνδρομή και η βοήθεια τεχνικού επίπεδου, τεχνικής φύσεως. Η πολιτική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πιο προηγμένη και αυτή η οποία παρέχει τους περισσότερους πόρους παγκοσμίως. Αλλά μέχρι ποιου σημείου μπορεί να υποφεληθούν κάποιες χώρες και επιχειρήσεις από αυτές τις συμφωνίες εάν δεν έχουν τα κατάλληλα στοιχεία στη διαθέσή τους. Τώρα, βελτίωση των υπαρχουσών ε, ε, συμφωνιών. Η εφαρμογή μια συμφωνία σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και τι μπορεί να βελτιωθεί. Το θέμα της παρουσίας των ε, δύο φύλων σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για πάρα πολύ ε, πολύπλοκες διαδικασίες. Θα πρέπει για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να κάνουμε αναθεώρηση του όλου συστήματος, γιατί μπαίνουν ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν βλέπουν το φως της γιατί δεν μπορούν να εφαρμοστούν και άρα δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ιαν Μαρίβιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για αυτή την πολύ λεπτομερή έκθεση. Θα ήθελα να εκφράσω λίγο την απογοητευσή μου. Πρόκειται για σημαντικές ε, συμφωνίες εμπορικές με πάρα πολύ επιφανειακές αναλύσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να επικρίνουμε αυτή την κατάσταση. Τελικά, ποιες είναι οι επιχειρήσεις που εποφελούνται από αυτές τις ε, συμφωνίες και ποιες είναι οι επιχειρήσεις που τελικά πλήττονται. Ξέρουμε ότι στην ε, περιοχή, σε άλλες περιοχές του κόσμου, Αλένα και στην Κορέα, υπήρξε επιδείνωση της κατάστασης, δηλαδή μειωμένη συμμετοχή σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Κύριε Πρόεδρε, καλό είναι να μας πει η Επιτροπή ότι όταν μιλάμε για προστασία των ειδών που απειλούνται, των φυτών της χλωρίδας της πανίδας, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτές οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει, έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, εάν ένας γιατρός μιλάει με τον ασθενή χωρίς όμως να υπάρξει καμία απόφαση για θεραπευτική αγωγή, δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι υπάρχει συζήτηση. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και αν αυτές οι συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες, συνεισφέρουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς το μετράμε, πώς μετράμε την πρόοδο. Συγκεκριμένα λοιπόν και εγώ θα ήθελα να έχω μια έκθεση που να δίνει λεπτομέρειες όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτών των επιτροπών. Πρόκειται ποτέ η Επιτροπή να μας υποβάλει κάτι τέτοιο. Οι εμπορικές συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες όπως ο Καναδάς, παραδείγματος χάρη, μειώθηκαν οι εισαγωγές από άλλες χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση καθόλου στον Καναδά. Γιατί παραδείγματος χάρη με το Βιετνάμ ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολύ καλή πρόσβαση μέσω του Βιετνάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και πριν απαντήσω συγκεκριμένα σε κάθε ερώτηση, θα ήθελα να σας πω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη Γενική μου Διεύθυνση, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τα σημεία που αφορούν την υλοποίηση. Το κάναμε αυτό από το 2015 και επίσης είναι σημαντικό η έμφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα να δίνεται περισσότερο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό τμήμα της δουλειάς μας αυτή την εποχή. Κοιτάξτε πόσος χρόνος δαπανάτε σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά την υλοποίηση, βεβαίως η υλοποίηση γίνεται όλο και πιο σημαντική όσο προχωράμε στη σύναψη της συμφωνίας. Βεβαίως συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό αντιστοιχεί και στη δική μας ανάλυση. Έχουμε όμως και ένα τρίτο σημείο. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις, έχουμε την υλοποίηση και έχουμε και ένα κομμάτι αμυντικών μηχανισμών. Επικαιροποίηση, ενημέρωση και προτάσεις όσον αφορά τον έλεγχο των επενδύσεων στις τρίτες χώρες. Μία συνεκτική πολιτική συμπεριλαμβάνει και τις τρεις αυτές και βεβαίως όλη αυτή η δουλειά εξελίσσεται, αλλά επαναλαμβάνω θα πρέπει να υπάρχει εξορροπημένη προσέγγιση και μέσω των τριών αυτών πτυχών της συμφωνίας. Κυρία Πλίστχαουτ, θα απαντήσω στην ερώτησή σας ότι έχουμε πολύ θετικά στοιχεία, έχετε δίκιο. Και για ποιο λόγο κάνουμε την έκθεση για να δείξουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις. Θέλουμε να προωθήσουμε αυτή την έκθεση όπου μπορούμε και στην ιστοσελίδα μας υπάρχει, αλλά και στα κράτη-μέλη και μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και θα συνεχίσουμε να την παρουσιάσουμε και το 2017 και έχουμε την εντύπωση ότι η έλλειψη συνειδητοποίησης, η έλλειψη γνώσης, γιατί όντως πολύ λίγοι γνωρίζουν για αυτές τις συμφωνίες, Προσπαθούμε να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αυξήσουμε την επικοινωνία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των εξαγωγών μέσω των ε, συστημάτων προτιμήσεως, ενημέρωση λοιπόν, πρόθεση των ε, εμπορικών συναλλαγών. Υπάρχουν κράτη, ε, κράτη-μέλη στα οποία αυτό γίνεται με πολύ περισσότερο ενθουσιασμό και σε άλλα που υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και δισταγμοί. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που εξηγεί ίσως λίγο το ότι τα θέματα αυτά δεν είναι πολύ γνωστά και δεν προκαλούν αρκετό ενδιαφέρον είναι και η περιπλοκότητα των μηχανισμών. Χρειάζομαι μια ειδική υπηρεσία, χρειάζομαι νομική βοήθεια. Αξίζει τον κόπο να προστρέξω σε αυτά εάν η διαφορά μεταξύ της σημερινής κατάστασης και των πλεονεκτημάτων που μου προσφέρει αυτή η συμφωνία είναι αρκετά, αν θέλετε, σημαντικά για να αξίζει τον κόπο. Εμείς προσφέρουμε εμπειρογνωμοσύνη, συμβουλή, στήριξη και θα ξεκινήσουμε και ένα πρόγραμμα το 2018 που θα απευθύνεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα των κανονισμών και των πιστοποιήσεων. Όταν εξάγεται ένα προϊόν, θα πρέπει βεβαίως να τηρούνται οι πολύ αυστηροί και συγκεκριμένοι κανόνες. Σήμερα, όπως ξέρετε, τα προϊόντα παράγονται σε πολλά στάδια και τελικά για να πιστοποιηθεί ένα προϊόν σαν ευρωπαϊκό, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ενσωμάτωσης της αξίας αυτού του προϊόντος στις διάφορες φάσεις της παραγωγής. Και θέλουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν και να κατανοήσουν αυτούς τους κανόνες. Κάποιος άλλος έκανε την ε, ερώτηση για τον οδικό χαρτί. Αυτό είναι μια νέα πρωτοβουλία, σχετικά νέα πρωτοβουλία για όλα τα νέα κράτη με τα οποία συνάπτουμε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και θέλουμε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος σε συνεργασία με τον λόγο κράτος μέλος για να είναι κατανοητό από τις δύο πλευρές τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης πρέπει να λάβουμε μέτρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί αυτό είναι μεγάλη βοήθεια στην υλοποίηση. Πρέπει επίσης να υπάρχει ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών σε όλα τα στάδια και τα κεφάλαια της ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου που τους αφορά. Οι συμφωνίες αυτές σίγουρα θα προκύψουν από τους αριθμούς που παρουσιάζουμε βλέπετε πόσο σημαντικές είναι είναι οι πληροφορίες που αφορούν τις ε, προελεύσεις, τη γεωγραφική προέλευση και ονομασίες. Ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν ε, είδη διατροφής, γεωργικά προϊόντα κτλ. Κυρία Πόστα, μιλήσατε για την ε, εκ των υστέρων αξιολόγηση και έλεγχο. Μέχρι τώρα οι προηγούμενες συμφωνίες ε, ελεύθερου εμπορίου αξιολογήθηκαν πριν το ξεκίνημα και κατόπιν έγινε αξιολόγηση συνεπειών κατά τη διάρκεια <clears throat> της συμφωνίας η κατεύθυνση, αν θέλετε, για τους διαπραγματευτές ε, δόθηκε μέσω αυτών που έκαναν αυτή την αξιολόγηση. Όσον αφορά την εκ των υστέρων ε, αξιολόγηση, θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα και παραπάνω από ένα χρόνο, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει να εκτιμηθεί, να αξιολογηθεί στην πράξη το αποτέλεσμα η συμφωνία. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο δηλαδή η αξιολόγηση να γίνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίηση της συμφωνίας και το πιο δύσκολο από όλα είναι η συλλογή των στοιχείων. Αυτό μου το λένε οι εμπειρογνώμονες από την αρχή. Η Eurostat έχει πληροφορίες με ως ένα συγκεκριμένο επίπεδο βέβαια. Αυτά τα στοιχεία που εμείς διαθέτουμε όταν θέλουμε να μπούμε σε συγκεκριμένες συμφωνίες που αφορούν ε, ατομικά τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο είδος ε, επιχειρήσεων, προσκρούμε πάντα στον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάποιων ε, δεδομένων Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη και ακόμα πιο δύσκολη είναι όταν προσπαθούμε να μαζέψουμε στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τις τρίτες χώρες. Μέσω των ε, συμφωνιών ε, ελεύθερου εμπορίου οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την άλλη πλευρά πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολο μπορούμε να τις αιτιολογήσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία. Μέσω της αξιολόγησης λοιπόν για την αποτελεσματικότητα μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου σίγουρα ίσως να μας δοθούν περισσότερες ευκαιρίες να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Και αυτό είναι ένα τομέα που σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί. Όσον αφορά την υλοποίηση, νομίζω μιλήσαμε γι' αυτό. Πιλωτικά προγράμματα. Αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σόλτς, η σχέση μεταξύ των FTAs, μεταξύ τους, η σύγκριση εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε θέσει τις βασικές προτεραιότητες. Οι επιχειρήσεις μας πρέπει να εποφελούνται. Αυτό είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Και... Βεβαίως. In the model that keeps prosperity in the European Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ευημερία και με απλό τρόπο μπορώ να πω ότι βεβαίως η πολιτική μας φιλοδοξία είναι πολύ μεγαλύτερη και θα θέλαμε να βελτιώσουμε την ε, ευημερία στις χώρες αυτές τις οποίες εξάγουμε. Βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους ε, στόχους μας, καλή διακυβέρνηση και σεβασμός βεβαίως των διεθνών προτύπων για την εργασία, για το περιβάλλον, όλα αυτά φυσικά και τα προάγουμε και θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των χωρών αυτών γενικότερα, όχι στον Καναδά βέβαια, αλλά στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στις γειτονικές χώρες. Γιατί βεβαίως υπάρχουν πολλά πολιτικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με αυτές τις συμφωνίες. Πώς γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση. τι αξιολογούμε την ανάπτυξη στις χώρες αυτές ως ένα βαθμό στο Μεξικό, στην Κολομβία. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα μας απασχολεί και θα πρέπει να αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε από κοινού. Τώρα, κάνατε και εσείς την ερώτηση για τη σύγκριση μεταξύ των Συμφωνιών Ελευθερίου Εμπορίου κάποιες τιμωρητικές ε, διατάξεις, κάτι που βεβαίως ξεπερνάει αυτή την έκθεση. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει για τα επόμενα χρόνια να μας απασχολήσει. Κύριε Φεράου, μιλήσατε για την ε, γεωργία. Ναι, υπάρχει πίεση του προϋπολογισμού και λιγότερα χρήματα θα διατίθενται για την γεωργία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνει η έκθεση μας δείχνουν ότι βεβαίως η γεωργία εποφελείται από τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, αλλά πολλές φορές δεν κατανέμονται ίσα και ομαλά τα πλεονεκτήματα από, αυτήν την, από αυτές τις συμφωνίες. και κάποιοι μπορεί να υποφεληθούν πολύ λίγο από μια τέτοια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Αν κοιτάξουμε όμως τη γεωργία γενικότερα και όχι μόνο σε σύγκριση με την κοινή αγροτική προητική, συνήθως μιλάμε για είδη διατροφής, για είδη διατροφής το οποία θέλει να αγοράσει, να εισάγει ο υπόλοιπος κόσμος. Και αν κοιτάξει κανείς επίσης τους αριθμούς, συγκεκριμένα βλέπει ότι τα υνοπνευματόδη, τα κρασιά, το ουίσκι είναι επίσης όσον αφορά την αξία αυτών των συμφωνιών ένας παράγοντας που σαφώς ε, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θετικό αποτέλεσμα των εμπορικών μας συναλλαγών με τις τρίτες χώρες. Έλλειψη γνώσης, έλλειψη κατανόησης ε, λέτε. Είναι περίπλοκα όμως τα συστήματα, μην το ξεχνάτε, και αυτό όχι μόνο για τις εξαγωγές μας, αλλά και για αυτούς που προσπαθούν να εξάγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. κυρία Μινάχ. Θα συμφωνήσω και ίσως εκπλαγείτε μαζί μου ότι πρόκειται για μια μάλλον ποσοτική ανάλυση και ότι δεν είναι αρκετά εις βάθος η ανάλυση μας. Ε, μιλήσατε για επιφανειακή έκθεση. Αλλά όπως σας είπα, πρόκειται για κάτι που φιλοδοξούμε να το βελτιώσουμε για τις επόμενες χρονιές. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ναι. Πρόεδρος, τέλεια. Είμαστε και στην ώρα μας. Απαντήσατε και σε όλες τις ερωτήσεις. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με το σημείο 6 και θα περάσουμε στο σημείο 7. Το 7 όμως είναι και κλεισμένων των θυρών. Κάνουμε λοιπόν μια μικρή διακοπή δύο λεπτών και όποιος ε, δεν ε, έχει το δικαίωμα να παραμείνει στην συνεδρίαση, παρακαλώ να εγκαταλείψει την αίθουσα.